Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω μία σύντομη ανακοίνωση σας κάνω εισαγωγικά. Πήρα ένα αίτημα της ομάδας του ΕΛΚΑ, της ομάδας των προεδρικών συμμαχίας των σωστών. και ελευθερών ε, της Δημοκρατίας και Ελευθερίας και Πρασίνων για καθορισμούς της επιτροπές και στις αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίας και αν δεν διαφωνήσει κανένας θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημέρας της διάταξης. Μια προφορική ερώτηση.